Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, περάστε στις θέσεις σας. Ξαναρχίζει η συνεδρίαση και θα λάβει το λόγο ο συνάδελφος Νέσμι Αλή. Έκθεση Ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στις 12 Ιουλίου 2016 οι κάτω χώρες υπέβαλαν αίτηση για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η αίτηση αυτή έχει να κάνει με απολύσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών. Αναφερόμαστε δηλαδή στην ε, στατιστική ονοματολογία ΝΕΙΣ ε, τομέα 47. Και αναφερόμαστε εδώ πέρα σε δύο περιοχές της ε, κατηγορίας ΝΑΤΣ επίπεδο 2, Ντρέντε και Οβερίζελ των κάτω χωρών. Το αίτημα αυτό ακολουθεί τους κανόνες ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με τους οποίους προβλέπεται ότι θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες πληρούνται. Ο αριθμός των εταιριών που έχουν πληγεί είναι συνολικά 6, ο συνολικός αριθμός των απολύσεων 1096, συνολικός αριθμός των ε, δικαιούχων 800 εργαζόμενοι είναι όλοι Ευρωπαίοι πίκο και περισσότεροι μάλιστα νέοι. Ο συνολικός προπολογισμός που προβλέπεται είναι 3.031.031 ευρώ και προβλέπεται εδώ πέρα συμμετοχή 60% με 1.818.750 ευρώ. Συμμετοχή 60% δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Λόγω της ε, οικονομικής ε, κρίσης λοιπόν που έπληξε και τη χώρα αυτή, προτείνεται να κινητοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απολύσεις αυτές, καθώς επίσης και η πάυση της εργασίας στον τομέα αυτό σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Πληρούνται λοιπόν οι σχετικές ε, προϋποθέσεις. Είναι επιλέξιμες οι αιτήσει αυτές και δεν αποτελούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας. Όλες οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως στόχο να καταφέρουμε να υπερβούμε τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από το κλείσιμο των καταστημάτων και των εργοστασίων αυτών. Όσον αφορά το αίτημα αυτό, θα ήθελα να σα πω ότι υπάρχει πρόταση ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώ επίση και πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση για δύο περιοχέ των κάτω χωρών, Ντρέντε και Οβερίζελ. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστούμε και εμεί. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ανταλλαγή απόψεων. Δεν ξέρω αν υπάρχει συνάδελφο που θα ήθελα να πάρει το λόγο. Ουδή μέχρι στιγμή. Ναι, συγγνώμη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ω κοιόδη εισηγητή για το ΕΛΚ να υποστηρίξω ότι το αίτημα αυτοκινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, γιατί τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ θα βοηθήσουν του 800 αυτού εργαζομένου 60% εξ αυτών είναι νέοι άνθρωποι κάτω των 25 ετών. Ειλικρινά λοιπόν υποστηρίζω την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα θέλει να πάρει το λόγο. Δεν νομίζω. Λοιπόν, οι τροπολογίες, αν θέλετε να καταθέσετε τροπολογίες, πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 9 Φεβρουαρίου. Ας περάσουμε τώρα στην χορήγηση εγγύησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης και δίνω ευθύς αμέσως το λόγο στην συνάδελφο Γκαρθιαμπάλ Ρουμπιάλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ενημερώσω τους ευρωβουλευτές, γιατί νομίζω ότι πότε ήταν προχτές, πήραμε ένα έγγραφο εργασίας για την εξωτερική επενδυτική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και είναι καλό να κοιτάξουμε λίγο αυτό το έγγραφο για να αναλύσουμε την κατάσταση και να καταλάβουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται και ποια ακριβώς είναι αυτή η εξωτερική επενδυτική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και να καταλάβουμε έτσι και την πρόταση της Επιτροπής και να έχουμε συζήτηση και να ακούσουμε τη θέση των διάφορων πολιτικών ομάδων και στη συνέχεια να καταλήξουμε σε έκθεση. Σήμερα λοιπόν θα σας πω ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία του εγγράφου αυτού εργασίας και μετά θα ακούσω, όπως σας είπα, τις πολιτικές ομάδες, γιατί με ενδιαφέρει να ξέρω περίπτωση πρόκειται. Το 2016, λοιπόν, το Σεπτέμβριο, η Επιτροπή πρότεινε μία αναθεώρηση τη εξωτερική αυτή εντολής τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για το 10% των δραστηριοτήτων της, της ΕΤΕΦ, και όπως πάντα ο προπολογισμό συμμετέχει με κάποια χρήματα, με εγγυήσει προ την ΕΤΕ συγκεκριμένα εγγυούμεθα για τις ενδεχόμενες ζημιές που μπορεί να προκύψουν από χρηματοδοτικές ε, δράσεις επενδύσεων που γίνονται στο εξωτερικό. Για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 υπήρχε η δυνατότητα για 30 δις εγγύηση. 27 έχουν ήδη ενεργοποιηθεί και μένουν και τρία τα οποία είναι σε... με ερωτηματικό ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν, μπορεί και όχι. Δηλαδή λειτουργεί λίγο πολύ όπως και το έτσι. Δεν τα έχουμε τα χρήματα 100%. Αυτό που κάνουμε είναι ότι εγγυούμεθα και το 2017, 18, 19 και 20, δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, περίπου 200 ε, δις άλλες χρονιές περισσότερα άλλες λιγότερα. Δίνουμε λοιπόν έτσι εγγύσει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να μπορεί να εκτελεί την εντολή της αυτή. Αυτό το Ταμείο Εγγύσεων χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό ετησίως, αλλά χρηματοδοτείται από τους τόκους από τα δάνεια επίσης. Ποια είναι η πρόταση λοιπόν τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, αναθεώρηση είναι μέρος του πακέτου αυτού του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου για την Αφρική και στόχος είναι να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τις κύριες αιτίες μετανάστευσης και να πετύχουμε έτσι τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Στις κύριες προτάσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι λέει, πρώτον θέτει έναν στόχο που είναι ακριβώς αυτός, να αντιμετωπίσουμε τις κυρίες αιτίες της μετανάστευσης. Ελευθερώνει αυτά τα 3 δισεκατομμύρια που όπως σας είπα πριν με έναν εμερωτηματικό, άρα λοιπόν από 27 δισεκατομμύρια πάμε στα 30 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η εντολή τώρα. Και επίσης προσθέτει και 2 δισεκατομμύρια 300 εκατομμύρια για να προσφέρει επιπλέον εγγύηση στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει αύξηση της εγγύησης από πλευράς ε, ε, του ευρωπαϊκού προπολογισμού κατά 114 εκατομμύρια. Θα πρέπει δηλαδή να πετύχουμε, αν μη τι άλλο, 182 εκατομμύρια συνολικά. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις που αναφέρονται για ένα νέο σύστημα δικτών, προκειμένου να μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα τα σχέδια αυτά, τα οποία απευθύνονται στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Υπάρχει και απαρίθμηση των χωρών που επιλέγονται. Υπάρχει κάποια ε, διαφορά με το Ιράν που μπαίνει τώρα στον κατάλογο. και υπάρχουν και δύο χώρες που βγαίνουν γιατί έχουν ένα επίπεδο ανάπτυξης αρκετά υψηλό. Προτείνει επίσης ενίσχυση της ευελιξίας, να μπορούμε δηλαδή από κάποιες εθνικές οροφές να μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα προς άλλες. Μέχρι ένα 20% μπορεί να προβλεφθεί αύξηση. Τώρα το Ταμείο Εγγύσεων, που είναι ακριβώς αυτό που αφορά το δικό μας προϋπολογισμό, που απορρέει από τη νέα συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, έχει σαν αποτέλεσμα νέα πηγή χρηματοδότησης. Πρόκειται για έσοδα από τα δάνεια αυτά επιπλέον. Η εγγύηση επίσης θα λειτουργήσει κάπως διαφορετικά. Έχουμε ένα 9% στο Ταμείο Εγγύησεων που βάζουμε για να εγγυθούμε την εξωτερική εντολή, αλλά υπάρχει και 1% ασφάλεια. Δηλαδή βάζουμε το 9% εμείς, αλλά το πρώτο 1% εσόδων που έρχεται μπαίνει στον προπολογισμό για να φτάσει το 10% και έτσι να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλά στον προπολογισμό θα κοστίσει 9%. Άλλη καινοτομία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι η χρηματοδότηση τη εγγύηση αυτή επιστρέφει για διαχείριση στα χέρια της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Δηλαδή η ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεν έχει πια τη διαχείριση τη εγγύηση αυτή. Αυτέ είναι οι προτάσει. Όπω βλέπετε υπάρχουν Όλα πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε και το πρώτο για το οποίο θα ήθελα την άποψη της Επιτροπής είναι κατά πόσο πιστεύετε πως η αύξηση που προτείνεται για την εγγύηση από πλευρά της Κομισιόν αρκεί από 27 δισεκατομμύρια φτάνουμε στα 31 και κάτι όπως είπαμε αλλά αν δούμε τα στοιχεία εκτέλεσης, χρήσης των κονδυλίων αυτών κάποια ε, δόθηκαν προκαταβολικά με την πρωτοβουλία για την νεολαία για παράδειγμα, όπου βάλαμε όλα τα χρήματα τα πρώτα χρόνια και μετά δεν μας μένει τίποτα. Και αλλού έχει γίνει το ίδιο. Και ζήτησαν οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ΕΤΕ να επικεντρωθεί περισσότερο στην Ουκρανία ή στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης και να δώσει προκαταβολικά τα χρήματα, οπότε τα τελευταία, χρώματα δεν, τα τελευταία χρόνια δεν θα υπάρχουν πια χρήματα για επενδύσεις. Υπάρχουν και αλλαγές που έχουν προκύψει στις χώρες. Υπάρχουν νέες χώρες που προκύπτουν και υπάρχουν και πολιτικές ε, αλλαγές. Κούβα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να συμμετάσχει και εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άρα χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις και σε άλλες χώρες. Ένα δεύτερο θέμα για το οποίο θέλω την άποψη των συναδέρφων είναι το εξή. Συμφωνούμε για την μεταφορά της διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χθε αναφερθήκαμε στο δημοσιονομικό κανονισμό και ένα από τα πράγματα που είπαμε ήταν η ιδέα αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει ενοποίηση των εγγυήσεων μέσα σε μία μόνο ε, γραμμή στον προπολογισμό. Γιατί έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και θα αποδοτήσουν καλύτερα τα χρήματά μας. Ήταν μια θετική πρόταση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε ρωτάω, θα υποφεληθούμε από αυτή την ευκαιρία για να μεταφέρουμε σιγά σιγά αυτή τη, σε αυτή την ενιαία ε, εγγύηση και τα χρήματα αυτά του εξωτερικού επενδυτικού σχεδίου. Συζητήσαμε χθε επίσης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτή η εξωτερική εντολή πώς θα συνδυαστεί με άλλους μηχανισμούς, είτε πρόκειται για τα καταπιστευτικά ταμεία, είτε για το blending, που υπήρχαν στον προϋπολογισμό και που κατά προτεραιότητα θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της μετανάστευσης στην Αφρική και άλλες πιο γειτονικέ μας χώρες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά όντως θα προσφέρουν μια προστιθέμενη αξία. Και το τελευταίο θέμα αλλά βλέπετε ότι εγώ στο έγγραφο εργασία μου βάζω ακόμα περισσότερε ερωτήσει. Πώ θα βελτιώσουμε την προβολή του έργου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ θα διασφαλίσουμε ότι οι δικαιούχοι όσοι αποδέχονται τελικά τα κονδύλια αυτά γνωρίζουν ότι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βελτιώσουμε τον έλεγχο και την ενημέρωση να γνωρίζουμε δηλαδή όλα τα στοιχεία ώστε να ξέρουμε τα κριτήρια που έχουμε βάλει, οι πολιτικές που έχουμε θέσει κατά προτεραιότητα όντω τηρούνται. Αυτά προς το παρόν από τη δικιά μου την πλευρά και περιμένω τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγητριά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα να απαντήσει παρακαλώ στις ερωτήσεις που έθεσε η εισηγητριά. Η κυρία Καρδιά Θαβάλα. Μπανζαμά Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλώς ορίζουμε το έργο του Κοινοβουλίου και της συζητήτριας. Μερικές παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, το μέγεθος της πρότασης. Αναμφίβολα, αν είχαμε μεγαλύτερο προπολογισμό, θα είχαμε καταφέρει περισσότερα. Ωστόσο, έπρεπε να το υπαγάγουμε στο τίτλο 4 του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου που έχει και τις περισσότερους περιορισμούς ως τίτλος. Η πρότασή μας αφορά μια πολύ σημαντική ανάπτυξη, αύξηση με μεγάλη προσπάθεια όχι μόνο να δώσουμε τα τρία δις επιπλέον, αλλά και το λέμε ότι δίνουμε και άλλα 2,3 δις Πράγμα το οποίο έχει άμεση επιπτώσει στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί σημαίνει ότι χρειαζόμαστε επιπλέον 300 εκατομμύρια στον προπολογισμό, εκ των οποίων τα, τωρινά, τα 35 στο τωρινό πουδουπού. Μπορεί να σας φαίνονται πολλά, αλλά στον τίτλο 4 είναι σημαντικό ποσό. Γιατί έχουν αδειάσει ούτως οι πίνοι τσέπες. Θα ήθελα επίση να διευκρινίσω, γιατί υπάρχουν και παρεξηγήσει και έχει γίνει και εκτεταμένη συζήτηση στο Συμβούλιο. Αυτό που προτείνει η Επιτροπή είναι για κάθε γεωγραφικό χώρο αύξηση και για τα ανατολικά. Δεν προτείνουμε να περιοριστούν τα ποσά. Καλύπτουμε λοιπόν ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση. Βέβαια η ΕΤΕ έχει περιλάβει την αλλαγή αυτή και προφανώς ε, θα πρέπει, γιατί δεν μπορεί να καλύψει ολόκληρη τη, όλες τις περιοχές με το ίδιο βήμα, με την ίδια ταχύτητα, έχει δηλαδή δαπανίσει περισσότερα στα ανατολικά και άρα θα πρέπει κάπως να προσαρμόσει την ε, προσέγγιση της, γιατί δεν είναι βιώσιμη αυτή η προσέγγιση μακροπρόθεσμα. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να διευκολύνουμε την ΕΤΕ να προχωρήσει βήμα το βήμα και έτσι να κάνει μια προσαρμογή του ίσταξους, να διατηρήσει δηλαδή το 10 με 20% για τα ανατολικά. Από την άλλη υπάρχουν και περιοχές, ζώνες όπως η Ρωσία, προς τις οποίες δεν υπάρχει καμία κινητικότητα και όσο δεν υπάρχει λόγος να τις υπολογίζουμε στην κατανομή. Διαχείριση πιστώσεων του Ταμείου Εγγύησεων, ε, μάλλον ενεργητικού Ταμείου Εγγύησεων, δεν είναι στην πρόταση βέβαια ακριβώ μέσα, αλλά θα πούμε ότι δεν έχουμε να προσάψουμε ή αδίποτε κατηγορία στην ΕΤΕ, αλλά έχουμε το εξής απλό ερώτημα να αντιμετωπίσουμε. Πληρώνουμε τέλη σχετικά υψηλά στην ΕΤΕ για να κάνει κάτι το οποίο θα μπορούσαμε εμείς να το έχουμε κάνει και δωρεάν. Επομένως, αποτελεί αυτό εξοικονόμηση τον ευρωπαϊκό προπολογισμό ή μήπω ε, τελικά αποτελεί κέρδο για τι ε, τράπεζε των κρατών. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε μόνο με την αγορά και πώληση securities χρηματοοικονομικών μέσων, χρηματοπιστωτικών μέσων για ε, τον προπολογισμό. Έτσι λοιπόν έχουμε εξοικονόμηση σε περίπτωση που τώρα λάβουμε εμεί ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Εάν όμως για κάθε μετοχή έχουμε χρέωση 11 ευρώ, στην περίοδο του Πουδουπού θα μπορούσαμε να έχουμε 66 εκατομμύρια σε δάνεια ή σε μακροοικονομική βοήθεια για ορισμένε χώρε ή σε δάνεια Euratom. Ε, Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα ποσά δεν αφορούν μόνο τις δράσεις της ΕΤΕ, αλλά πολύ ευρύτερη κατανομή. Και γι' αυτό λοιπόν χωρίς να θέλουμε κανένα να περιορίσουμε και καμία δραστηριότητα, μπορούμε τώρα να διαθέτουμε περισσότερα χρήματα για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό από ότι μπορεί να προσφέρει η ΕΤΕ χωρίς να θέλουμε να την επικρίνουμε. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Όταν έχουμε δική μας τράπεζα, γιατί να πάμε να καταβάλουμε τα τέλη και τις χρεώσεις ενός εξωτερικού τραπεζίτη. Έτσι, πολύ πιο φθηνό. Τελευταία παρατήρηση. Κοιτάξαμε τον κατάλογο των επιλέξιμων κρατών και τον μειώσαμε ουσιαστικά γιατί περιελάμβανε και χώρες που δεν είχαν πλέον θέση καθώς ε, όλες από αυτές έχουν εισόδημα πολλές φορές ακόμη και υψηλότερο από πολλών κρατών μελών. Φερρυπίν, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ισλανδία, Ισραήλ, Επομένως, στις χώρες υψηλού εισοδήματος, τις βγάζουμε από τον κατάλογο, δεν έχει λόγο να τις κρατάμε. Το Συμβούλιο έχει συμπληρώσει από τον κατάλογο αυτόν μία πρόταση, μία χώρα, χωρίς εμείς να το εγκρίνουμε και είναι η Ταϊβάν αυτή. Η Επιτροπή προτείνει να βγάλουμε το Χονγκ Κόνγκ και το Μακάο. Κάπως λησμονήθηκε όμως η Ταϊβάν, πάντως και για αυτήν ισχύουν τα ίδια επιχειρήματα μία χώρα και μία μόνο χώρα προτείνουμε να συμπληρωθεί στον κατάλογο πιθανώς επιλέξιμων χωρών το Ιράν. Το Ιράν, Αϊράν όπως λέει ο μιλητής, δεν ξέρουμε, δεν σημαίνει ότι θα είναι ε, αυθορή επιλέξιμο. Θα δούμε αν θα καταστεί επιλέξιμο με βάση κάτι εξουσιοδότηση πράξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ΑΕΡΑΝ. Και βεβαίω θα έχουν δικαίωμα και άρνηση κυρία στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εάν αποφασίσουν να μην υποστηρίξουν την επιλεξιμότητα του ΑΕΡΑΝ όταν έρθει η ώρα. Θα σταματήσω εδώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Μα προκαλεί φοβερή έκπληξη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δανειοδοτεί τελικά τη Σιγκαπούρη. Πραγματικά υπάρχει εδώ πέρα κάποιος οδικός χάρτης, ξέρουμε πού πηγαίνουμε, υπάρχει κάποιο όραμα στρατηγικό όσον αφορά τα δάνεια αυτά, δίνουμε δεξιά και αριστερά εμείς δάνεια απλόχερα τελικά. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω και θα ήθελα να καταλάβω τελικά τι συμβαίνει και αν υπάρχει κάποια λογική μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινήσεις αυτές. Ενδεχομένως να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι υπόλοιποι ομιλητές παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Λέει ο κύριος Μουρεζάν. Χαιρετίζω και εγώ την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει την εξωτερική δανειοδοτική εντολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θεωρώ ότι η εξωτερική αυτή δανειοδοτική εντολή πρέπει όντως να χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στην άμεση γειτονία μας. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να γίνουν ιδίω στο πλαίσιο της αστάθειας που βλέπουμε στα ανατολικά τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει πάση θυσία να υποστηρίξουμε χώρες όπως η Ουκρανία προκειμένου να καταφέρουν να έχουν πιο σταθερές δημοκρατικές δομές, πιο σταθερή οικονομία και θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στις χώρες της ανατολικής και νότιας γειτονίας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που έχουμε για τους διαθέσιμους πόρους μας. Όσον αφορά καταρχάς τον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών, πολύ σωστά αποκλείουμε πλέον από τον κατάλογο αυτό αναπτυγμένες χώρες και οι οποίες δεν χρειάζονται άμεσα δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αναφέρομαι προφανώς τη Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, τη Ισλανδία και τις υπόλοιπες χώρες που ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ θετικό που προσθέτουμε πλέον το Ιράν στις δυνάμει επιλέξιμες χώρες. Αυτό όμως από μόνο του δεν σημαίνει ότι αυτόματα το Ιράν θα αρχίσει να λαμβάνει δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βραχυπρόθεσμα. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την τη της χώρας αυτής. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν απαραίτητε δομέ προκειμένου και στην περίπτωση του Ιράν αλλά και στην περίπτωση των υπόλοιπων χωρών όντω τα χρήματα να πηγαίνουν στου άμεσου αποδέκτε, μικρομεσαίε επιχειρήσει και γενικά στου ανθρώπου εκείνου που χρειάζονται την οικονομική υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Α συμπεριλάβουμε λοιπόν και το Ιράν στον κατάλογο αυτό αλλά α μην το χρηματοδοτήσουμε και από την πρώτη μέρα. Όσον αφορά τώρα τα όσα μας είπε η συγγήτρια για τις προτάσεις αύξησης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν όντως μας βρίσκουν σύμφωνους, πώς έχει η κατάσταση επί του παρόντος. Βλέπουμε ότι ένα 46% της εξωτερικής ανεδοτικής εντολής της ΕΤΕΠ ήδη χρησιμοποιήθηκε μέχρι τα τέλη του 2016 και βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο κρίσιμη αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Γειτονία. Ένα 84% των ποσών που είχαν δοθεί χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τα τέλη του 2016. Και για ποιο λόγο η δανειοδοτική δράση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ήταν ιδιαίτερη, ιδιαίτερα έντονη όσον αφορά την Ουκρανία. Για την Ανατολική λοιπόν γειτονία η αύξηση από 4,8 δισεκατομμύρια ως 6 δισεκατομμύρια δεν αρκεί. Αν συνεχιστεί η τάση αυτή απορρόφηση πόρων ή ανάγκη, ανάγκης νέων πόρων στην Ουκρανία και γενικότερα στην Ανατολική γειτονία, μέχρι τα μέσα του 2018 θα έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμοι πόροι. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη χρηματοδοτική υποστήριξη της ε, περιοχής αυτής ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ φοβάμαι ότι είτε θα σταματήσει η δανειοδότηση, θα είμαστε σε θέση να δίνουμε μικρότερα τελικά δάνεια αν δεν αυξηθούν οι πόροι. Πρέπει λοιπόν να αυξηθεί καταρχάς η δυνατότητα χρησιμοποίησης της ρήτρα ε, ευελιξία να περάσει αυτή από 10% στο 20% έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μπορέσει τελικά να δώσει προτεραιότητα στις χώρες εκείνες, στις περιοχές εκείνες που έχουν στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η άμεση νότια γειτονία και ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα, αν θέλετε, ή θα πρέπει να βρίσκονται ψηλότερα στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων από ό,τι χώρες της ε, Νοτιοαμερικής ή τη ε, έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία λοιπόν και α χρησιμοποιήσουμε του πόρου για τι πιο σημαντικέ περιοχέ εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου τελικά οι δεσμεύσει μα προ τι χώρε αυτέ θα πρέπει να διακοπούν ή δεν θα μπορέσουμε να τι στηρίσουμε. Για να απαντήσω και στα ερωτήματα τη εισηγήτρια, το να καταφέρουμε να φτάσουμε τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το ελάχιστο που μπορούμε να απαιτήσουμε ιδανικά προκειμένου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μπορεί να ολοκληρώσει την εντολή της, θα πρέπει να είχαμε 38 δισεκατομμύρια. Η αύξηση να φτάνε τα 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να δούμε βέβαια και ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι. Η άποψή μου πάντως είναι ότι η αύξηση στα 35-36 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η ελάχιστη αύξηση που θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεχίσει τι δραστηριότητε της. Ένα ερώτημα να θέσω κι εγώ όσον αφορά την Ανατολική γειτονία και πιο συγκεκριμένα την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πώς θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη χώρα αυτή, την Ουκρανία, δεδομένου του ότι ε, εκεί πέρα δόθηκαν τα μεγαλύτερα ποσά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κινδυνεύουμε να σταματήσουμε τη χρηματοδοτική υποστήριξη της χώρας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έκανε προς την Ουκρανία και ποιες ήταν οι επιπτώσεις για τις υπόλοιπες χώρες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το μεγαλύτερο τμήμα της χρηματοδότησής μας στα πλαίσια της πολιτικής ανατολικής γειτονίας πηγαίνει στην Ουκρανία. Τι θα γίνει όμως με τις υπόλοιπες χώρες όπως η Γεωργία, η Μολδαβία που και αυτές περιμένουν χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή έχουν υπογράψει και συμφωνίες σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. πριν ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την ΕΤΕ να απαντήσουν, ο κύριος Μπέγκε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω στο όσα υπόθηκαν μόλις τώρα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν εισηγητής από πλευρά του Κοινοβούλου, αλλά ήμουνα παρόν εγώ ως βουλευτής όταν έγιναν την πραγματεύση της πρώτες εντολές για εξωτερικές δράσεις της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Και έχουμε δει τα τελευταία χρόνια την ΕΤΕ να αναλαμβάνει μια σειρά από συγκεκριμένε επιλογές με ευθύνη βέβαια της διοίκησής της γιατί βέβαια οι εγγυήσει ποτέ σχεδόν δεν υιοθετήθηκαν ως προσέγγιση. Αυτό που είπε η συνάδελφος συγγήτρια είναι πολύ σημαντικό ότι η συμπλήρωση του εργαλείου αυτού για την εξωτερική εντολή δεν μπορεί να εξεταστεί με μονομένα δεδομένης της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε στη γειτονία μας, στα Ανατολικά, στη Μέση Ανατολή, στα Νότια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια άκρος δύσκολη κατάσταση και μάλιστα κράτη κατεστραμμένα πολύ συχνά, μας γεννούν ανησυχίες και για την ανθεκτικότητα στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ως εκ τούτου εγείρεται το ερώτημα, τι έχουμε κάνει ή τι έχουμε παραλείψει ενδεχομένω στο παρελθόν για τη σταθεροποίηση της γειτονίας αυτής την περί, ε, περιοχή. Εγώ δεν λέω ότι πάντα χρειάζεται ένα νέο εργαλείο και ότι πάντα αυτό θα αποτελεί τη λύση γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε και τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρουν τα υφιστάμενα προγράμματα για τη γειτονία. Γι' αυτό εγώ δεν θα κοίταγα μόνο την τεχνική προσέγγιση, χρηματοοικονομικά τεχνική προσέγγιση, αλλά την πολιτική προσέγγιση πώς μπορούν να αλλάξουν ε, και τι είδους συνοχή μπορεί να προσφέρουν, πώς να φέρουν αλλαγές δηλαδή, αλλά και τι είδους συνοχή μπορεί να προσφέρουν τα εργαλεία αυτά με βάση τη στόχευσή μας και εκεί βέβαια γύρεται και το ερώτημα του ύψους των εγγύσεων που θέλουμε να δώσουμε. Γι' αυτό εγώ θα προτιμούσα μια ολιστική προσέγγιση για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του εάν και πώς θα καταφέρουμε τα αποτελέσματα που έχουμε ήδη από το παρελθόν προσδιορίσει. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι το εξή. Και εδώ δεν θα συμφωνήσω καθόλου με τον Ζίκφριτ. Είμαι μέλος της αντιπροσωπείας για τη σχέση με την Χιλή και την Eurolat. Και στην ομάδα ε, επιτήρησης monitoring για την Κεντρική Αμερική. Όντω δεν πρέπει ορισμένε χώρες να μπουν στον κατάλογο αυτό. Είναι σωστό το ότι δεν έχουν μπει. Αλλά η στρατηγική πολιτική και οικονομικοστρατηγική θεώρηση της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε τώρα και με την εκλογή του Τραμπ και την καταγγελία της, ε, την διακοπή των διαπραγματεύσεων ε, της ε, συμφωνίας για τις σχέσεις εμπορικές με τις χώρες του ειρηνικού από πλευρά του Τραμπ δείχνει ότι οι χώρες αυτές βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και θα βρεθούν σε ακόμη πιο δύσκολη και άρα έχουμε εμείς και μεγάλη πολιτική ευθύνη. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να κοιτούμε μόνο την άμεση γειτονία μας Ανατολή, Μέση Ανατολή, Νότος της Ευρώπης. Θα πρέπει να αναλάβουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο τις ευθύνες μας και να ε, κινηθούμε προς τις κατευθύνσεις αυτές. Γι' αυτό προς τον Πρόεδρο απευθύνω και την έκκληση να αξιοποιηθεί, προς όλους μάλλον, να αξιοποιηθεί η περίοδος ε, μέχρι την κατάθεση των τροπολογιών που έχουμε για την προθεσμία μέχρι την κατάθεση των τροπολογιών για να κάνουμε και μια ακρόαση ενδεχομένως κύριε Πρόεδρε να μπορέσουμε να δούμε τους ειδικού που θα μας δώσουν περισσότερα στοιχεία. Λοιπόν ευελιξία ναι θα συμφωνήσω, περισσότερη ευελιξία όμως δεν μπορεί να σημαίνει ή να οδηγήσει στο να παραγνωριστεί αυτό το οποίο χτες συζητήσαμε ακόμη, δηλαδή τη δυνατότητα ε, εμπλοκής του Κοινοβουλίου σε αυτές τις διαδικασίες, τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Και σε αυτό πρέπει ξεκάθαρα να αποστείλει και τα μηνύματα της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμμετοχή μας στα εργαλεία αυτά που θα ε, διαπραγματευτεί τους επόμενους μήνες. Άλλος κανείς? Πρόεδρος. Λοιπόν, με αυτό το έγγραφο εργασίας πιστεύω ότι έχουμε μία συζήτηση που είναι ουσιαστικότατη, κεφαλαιόδου σημασίας. Γιατί οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε έχουν να κάνουν με την ίδια την στρατηγική, το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να ξέρω πράγματι ποιος είναι ο χάρτης πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από αυτόν. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με γεωπολιτικά ζητήματα. Όταν βλέπω ότι δίνουμε σε κινέζικες περιφέρειες δάνεια, ενώ η Κίνα μας δανείζει, θα ήθελα να καταλάβω ποια είναι η λογική του πράγματος. Είναι γιατί, για να βοηθήσουμε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αλλά αξίζει νομίζω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση ουσίας για τη θέση που θέλουμε να έχει η Ευρώπη στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. και να δούμε ποια είναι η θέση της ΕΤΕ και των εγγύσεων που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ΕΤΕ. Πέρα από τα εξαιρετικά που μας είπε η συγγήτρια και τις παρεμβάσεις των συναδέρφων, παραμένει κεφαλαιόδου σημασία το ζήτημα που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πραγματικής συζήτησης στην Ολομέλεια, γιατί είναι κάτι που αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Καλώς. Μια κυρία Σέλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω, λέει η κυρία Νεριάντα, πως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την σταθερότητα και την ανάπτυξη που χρειάζονται επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές, στην εκπαίδευση, στην υγεία. Είναι πολύ σημαντικό να τα πετύχουμε όλα αυτά και βέβαια και διαφάνεια και λογοδεσία. Πήρα μια φωτογραφία τον ε, μηχανισμό των χρηματοδοτικών που εξετάζαμε χτες στην, ε, στο εργαστήριο που είχαμε για τον γαλαξία τέτοιων μηχανισμών και όντως πρόκειται για χάος. Πώς θα έχει πρόσβαση ο κόσμος σε αυτά, εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω, οπότε πώς θα καταλάβει ο κόσμος όταν μιλάμε λοιπόν για διαφάνεια και για λογοδοσία, πώς θα τα πετύχουμε όταν εκπονούμε έγγραφα τόσο περίπλοκα τόσο δύσκολα κατανοητά, πώς θέλετε να καταλαβαίνει ο κόσμος. Φυσικά και πρέπει να στηρίζουμε τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να δούμε και τις κοινωνικές επιχειρήσεις, γιατί η κοινότητα πρέπει να ενισχυθεί. Για να πετύχουμε την, την βιωσιμότητα φυσικά και χρειάζεται σταθερότητα και ανάπτυξη. Και φοβάμαι ότι κάνουμε ανάποδα τα πράγματα, από πάνω προς τα κάτω και όχι από κάτω προς τα πάνω. Επίσης, η ΕΤΕ δεν αντιμετωπίζει και τα ζητήματα των μικρών δανείων. Κάτι το οποίο όμως είναι πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε η ΕΤΕ να μην έχει ενδιάμεσους, γιατί τελικά καταλήγουμε να έχουμε πάρα πολλά επίπεδα γραφειοκρατίας υπάρχει η διευκόλυνση των πιστώσεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια άμεση σχέση και λιγότερο γραφειοκρατική για να παίρνουν χρήματα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε θα ήθελα η ΕΤΕ να αποκτήσει κάποιο μηχανισμό που θα την καταστήσει λιγότερο γραφειοκρατική για να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις κοινωνικές εταιρείες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Δεν βλέπω να ζητάει κανένας άλλος το λόγο. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε από τον κύριο Μπέρν της ΕΤΕ να μας εξηγήσει πώς γίνονται τα πράγματα εκεί. Πώς γίνεται η αίτηση για δάνεια από επιχειρήσεις, από κρατικούς φορείς, ποιος είναι ο μηχανισμός. Και τελικά ποιο είναι, ποιος είναι ο χάρτης πορείας που έχετε, ποιος τον ε, εκπονεί. Είναι οι πολιτικές αρχές, είναι το διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Δεν θα σχολιάσω αυτά που ακούσαμε στην αρχή, είναι πολύ τεχνικά, είναι προτάσεις που γίνονται από διάφορους παράγοντες και θα έπρεπε να εξεταστούν σε μια ανεξάρτητη έρευνα. Αλλά, ναι, όντως έχουμε ε, πολύ καλές επιδόσεις με αποτέλεσμα να μπορούμε να δώσουμε τα 700 εκατομμύρια δάνεια. Όμως θα ήθελα να ε, αναφερθώ στον κατάλογο αποκλεισμού που αναφερθήκατε. Καμία από αυτές τις χώρες δεν έχουν χρησιμοποιήσει τον εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο για πολύ καιρό. Ακριβώς γιατί έχουμε μία πολιτική χορήγηση κονδυλίων όπου ακόμα και χώρες όπως η Τουρκία που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε άλλη εγγύηση, χρησιμοποιούμε την δικιά μας εγγύηση, αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία. Πέρυσι βασιστήκαμε στους ιδίους κινδύνους και όχι σε αυτό το Ταμείο Εγγυήσεων, επειδή ακριβώς έχουμε μια τέτοια πολιτική χορήγησης δανείων δεν δανείζουμε στη Σιγκαπούρη, στη Νότια Κορέα και τα λοιπά από το εξωτερικό επενδυτικό μας σχέδιο. Το άλλο που ρωτήσατε είναι ποια είναι η στρατηγική μας. Η ΕΤΕ είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε η στρατηγική μας είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χαράσεται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι το παράδειγμα των ανατολικών περιοχών όπου αναφέρθηκαν πολλοί. Μας ζητήθηκε να αυξήσουμε τον δανεισμό μας προς αυτές τις χώρες κατά 3 δισεκατομμύρια. Δεν ήταν επιπλέον ε, πληρωμές, ήταν η ανταπόκρισή μας στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βάσει των οποίων λειτουργούμε. Ήταν η εντολή που πήραμε. Ο δανεισμός αυτός λοιπόν βάσει των ευρωπαϊκών πολιτικών χορηγήθηκε, μας ζητήθηκε να αυξηθεί όπως είπαμε κατά τρία δις, εκτός από την εγγύηση. Γι' αυτό και τώρα προβλέπουμε αύξηση. Σίγουρα οι ανατολικές περιοχές δεν καλύπτουν τα 3 δισεκατομμύρια. Θα πάμε κάτω από τα όρια δανεισμού που υποστηρίζαμε πριν από το πακέτο για την Ουκρανία. Όμως με τα όρια έτσι όπως έχουν τώρα βάσει της νομοθεσίας, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ε, πια δανεισμό στην Ουκρανία στα επίπεδα ε, που είχαμε, ούτε και ποθενά αλλού στις ανατολικές ε, περιοχές, ακριβώς εξαιτίας των κονδυλίων που εξαντλήθηκαν πέρυσι. Συνεπώς, για να παραμείνουμε στα όρια των εγγύσεων και στην περιοχή αυτή είναι δύσκολος ο δανεισμός. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Ο πολιτικός κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, όπως καταλαβαίνετε. Θα μειώσουμε το δανεισμό ε, φέτος, λίγο του χρόνου και μετά θα σταματήσουμε. Αν μείνουν τα όρια σημαίνει ότι σταματάμε το δανεισμό στην Ουκρανία αλλά και στις άλλες χώρες της περιοχής. Πάντα για τη στρατηγική εννοείται ότι δεν δανείζουμε στη Ρωσία και ότι υπάρχει κανένα τέτοιο σχέδιο για δανεισμό στη Ρωσία βάσει των πολιτικών εντολών που λαμβάνουμε. Για την ευελιξία τώρα. Στην νομοθεσία φυσικά και το εκτιμάμε ιδιαίτερα πώς να το πω, από μια το θέλουμε, απ' την άλλη πιέζουμε με ευελιξία την ΕΤΕ για να τα καταφέρει εκεί που είναι δύσκολο. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να πούνε τι θέλουν να στηρίξει η τραπεζά τους. Τέλος, για τη στρατηγική μας. Κίνα, ναι, δανείσαμε, αλλά μόνο στα πλαίσια της κλιματικής δράσης, που είναι υψηλή προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθούμε λοιπόν τις καταφεδρίες ε, αμέσως. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο αγαθό το περιβάλλον, οπότε η στήριξή μας πηγαίνει παντού. Και η Κίνα ε, έχει βέβαια ορυκτά καύσιμα που καίει, οπότε αν θέλουμε να βοηθήσουμε στο τομέα του περιβάλλοντος, τότε πρέπει να βοηθήσουμε την Κίνα να αλλάξει. Πρόεδρος διακόπτη. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Λέμε δανείζουμε στην Κίνα για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Δανείζουμε λοιπόν στην Κίνα ως κράτος ή δανείζουμε σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν ε, στην ε, Κίνα σε διάφορες εργασίες και που είναι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σε ποιον δανείζουμε ακριβώς στην Κίνα. Στην περίπτωση αυτή στον ιδιωτικό τομέα. Ο δανεισμός είναι κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επίσης Διακόπτη πάλι ο πρόεδρο, αυτές οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι κινέζικες ή ευρωπαϊκές. Πρόκειται για το διεθνές επίπεδο, δηλαδή διεθνείς επιχειρήσεις. Αυτές ζητούν. Και αυτές στηρίζουν τα προγράμματα που θέλουμε και εμείς να χρηματοδοτήσουμε. Ακολουθούμε, όπως σας είπα, τις διαδικασίες των διαγωνισμών, διεθνών διαγωνισμών και βάσει αυτών δανείζουμε. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι γίνεται διεθνής διαγωνισμός ή καλύτεροι, καλύτερες επιχειρήσει που φαίνεται ότι θα προσφέρουν, ξέρω εγώ, θα φτιάξουν γεννήτριε ή οτιδήποτε άλλο, παίρνουν τα δάνεια. Πολλές φορές πρόκειται για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά πρόκειται για διεθνείς διαγωνισμούς, πρόεδρος. Και παρεμβαίνουμε γιατί, γιατί αυτοί που κέρδισαν το διαγωνισμό είναι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που βοηθάμε. Αν δεν είναι ευρωπαϊκές, τελικά δεν δίνουμε δανεισμό. Αυτό θέλω να μου διευκρινίσετε. και σε μη ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δανείζουμε. Ακριβώς γιατί αυτή είναι η ευρωπαϊκή πολιτική. Να στηρίξουμε το ελεύθερο εμπόριο ανοιχτά και βάσει αυτής της πολιτικής κάνουμε τους διεθνείς διαγωνισμούς και όποιος κερδίσει. Δεν θα στηρίζαμε τοπικά ε, η ανδική κυβέρνηση για παράδειγμα θέλει να φτιάξει ε, συμμετέχουν μόνο ειδικέ ε, επιχειρήσεις, εμείς δεν θα προσφέρουμε δανεισμό τότε. Γιατί θέλουμε να υπάρχει ανοιχτός διαγωνισμός. Αν όμως υπήρχε μια επιχείρηση από το Μεξικό που μπορούσε να προσφέρει καλύτερο εξοπλισμό για ένα ολικό πάρκο, τότε ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πολιτική, ό,τι λέει η ευρωπαϊκή πολιτική που λέει σε αυτή την περίπτωση ανοιχτή διαγωνισμή. Και αν δείτε το αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής, πολλές φορές τις περισσότερες, θα έλεγα, κερδίζουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Απαντάω έτσι στην ερώτησή σας. Πρόεδρος, δηλαδή, για να καταλαβόταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χρειάζεται χρήματα για να χρηματοδοτήσει οι Κινέζοι μπορεί να συμμετάσχουν σε δάνεια της, ε, που προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία προφανώς πρέπει να έχει χρήματα, για να χρηματοδοτήσει μετά με δάνεια την Κίνα πάλι. Ναι, 100% έτσι κι αλλιώς εμείς δεν δανειοδοτούμε τίποτα. Θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς συγχρηματοδότηση. Έτσι διασφαλίζουμε και την έλευση και άλλων πηγών χρηματοδότησης. Συμμετέχουμε όσο χρειάζεται ώστε να λάβει χώρα ένα έργο. Μπορεί να είναι 20% και το 80% να το προσφέρουν άλλοι. Για μας είναι πολύ καλό αυτό. Σημαίνει αυτό στο κλίμα. Θα μπορούσε να πρόκειται για Κινέζους επενδυτές που συμμετέχουν επίσης ή για άλλους Ευρωπαίους ε, επενδυτές. Τι άλλο. Νομίζω ότι έχω απαντήσει, αλλά ναι, κάτι ακόμα. Ρωτήσατε τρέχον σύστημα εγγύσεων επιτρέπει συνεχή δανεισμό στα σημερινά επίπεδα. Όχι, διότι έχουμε χρησιμοποιήσει ήδη τα όρια εγγύσεων και έχουμε 60% μείωση του δανεισμού στις ανατολικές περιοχές. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε αμέσως, έτσι κι υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία αν η νομοθεσία παραμείνει ως έχει, πρέπει να επιβραδύνουμε. Και μετά το 2018 δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε το δανεισμό στις ανατολικές περιοχές. Η τελευταία ερώτηση ήταν για αυτή την πληθώρα χρηματοδοτικών μηχανισμών, τον Γαλαξία. Υπάρχουν πράγματι πολύ διαφορετικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την εκπόνηση πολιτικών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΤΕ, εφόσον είμαστε Ευρωπαϊκή Τράπεζα, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να υπάρχει συμπληρωματικότητα και οι μηχανισμοί αυτοί να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρησιμοποιούμε και άλλους μηχανισμούς. Υπάρχουν οι διευκολύνσεις στις χώρες ΑΚΕ, Επίσης υπάρχουν τα επενδυτικά ταμεία, οι ίδιοι πόροι των χωρών και όλα αυτά μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε διάφορες προκλήσεις. Και βάσει αυτής της λογικής θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και τις αιτίες της μετανάστευσης. Για τις μικρομεσαίες τώρα που ρωτήσατε. Συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα. Και το κάνουμε με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι υποστηρίζουμε το, την οικονομική ανάπτυξη. Γιατί αυτό που χρειάζεται σε διάφορες χώρες είναι ένας ε, γερός οικονομικός ε, κλάδος, χρηματοπιστωτικός. Και αυτόν τον ενισχύουμε πολλές φορές. Και ο άλλος τρόπος είναι προγράμματα με μικροπιστώσεις στην υποσαχάρια Αφρική, για παράδειγμα, 500 εκατομμύρια ή με τους αδέρφους της Κομισιόν και της χώρες μέλη το κάνουμε και για τη Βόρεια Αφρική και τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάντως συμφωνώ με τον Πρόεδρο ότι χρειάζεται μια συζήτηση ουσίας προκειμένου οι μηχανισμοί για την ευρωπαϊκή ε, ανάπτυξη να διέπονται από συνοχή και να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένη γραμμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ευχαριστούμε για όλε αυτέ τι διευκρινήσει. όντω θα πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη συζήτηση, ένα εργαστήριο ενδεχομένω ή μια ακρόαση για όλα αυτά τα ζητήματα χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ άλλε περιοχέ και να δούμε αν υπάρχει πραγματικά ένα στρατηγικό όραμα κατά την δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλες περιοχές. Δεν ξέρω αν ο κύριος Αντζέλ, εξ νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να κάνω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις, κάποια σχόλια, καταρχάς ε, όσον αφορά το asset management, τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού. Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έχει απόλυτα δίκιο. Έχει καταφέρει η τράπεζα αυτή να δημιουργήσει κέρδος και έσοδα και αυτό γίνεται επίσης και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι τα τέλη τα οποία εμείς πληρώνουμε προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα καθαρό κόστος το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε αναλάβει εμείς εσωτερικά ή να είχαμε γλιτώσει ουσιαστικά. Όσον αφορά τώρα τα συνολικά ποσά τα οποία δίνονται, σαφώς θα πρέπει να γίνει μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων. δεν αποτελεί προτεραιότητα για μας κάθε περιοχή του κόσμου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερθήκαμε στην ανατολική και νότια γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως πρέπει να επικεντρωθούμε στις χώρες αυτές. Πρέπει να ασχοληθούμε επίσης με την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Οι πρόσφυγες δεν έρχονται από την Κίνα και την Βραζιλία. Ας είμαστε ειλικρινείς. Χρειαζόμαστε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εκμεταλλευτεί κάθε δυνατή ευκαιρία προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιεί εφιώς, αν θέλετε, αυτή την περαιτέρω ευελιξία που εμείς προτείνουμε να διατηρηθεί για αυτούς, η οποία είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να ισχύει αυτή η ρήτρα ευελιξίας. Πέρα από αυτό όμως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επικεντρώνεται και σε περιοχές οι οποίες μπορεί να μην αποτελούν άμεση προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκεί πέρα θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να χρησιμοποιεί τους δικούς της μηχανισμούς εγγύσεων. Και αναφέρομαι στη δανειοδότηση της ε, Κίνα ή άλλων περιοχών. Πρέπει να χρησιμοποιεί και στι περιοχές αυτές που δεν αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι. Όταν χρηματοδοτεί την Κίνα, χρησιμοποιήσει το δικό της σύστημα εγγύσεων και τους δικούς της ιδίου πόρου το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ανοιχτό αν θέλετε ATM το οποίο απλόχερα και γενναιόδωρα θα χρηματοδοτεί κάθε περιοχή του κόσμου. Μακάρι να ήταν έτσι. Μακάρι να μπορούσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτεί απλόχερα και 100 φορές περισσότερο από το κάνει τώρα. Αλλά στην πράξη δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε λευκή επιταγή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή ένα ανοιχτό σύστημα εγγύσεων. Μακάρι να μπορούσαμε. Το θέμα είναι ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι και πώς αυτοί ε, ρυθμίζονται στα πλαίσια του ε, δημοσιονομικού πλαισίου που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι να είχαμε ανεξάρτητους πόρους, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι οι πόροι όλο και μειώνονται και πολλές φορές δεν έχουμε καν πόρους για να συνεχίσουμε την αδειοδότηση περιοχών που είχαμε δανειοδοτήσει στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε πολλές φορές στις δεσμεύσεις μας. Όταν ο νομοθέτης ψήφισε τον ELM, είχαμε πει ότι θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε με 3 δισεκατομμύρια. Εμείς δώσαμε πολύ περισσότερα όμως. 4-5 δισεκατομμύρια επιπλέον. Δεν ξέρω όμως πώς μπορούμε αυτή τη στιγμή να προσθέσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα και να ανταποκριθούμε στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Προφανώς θα αντιμετωπίσει ΕΤΕ προβλήματα στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Είναι δικό τους όμως αυτό καθήκον και πρέπει να το καλύψουνε αλλά αυτή τη στιγμή ε, ως εκδιαμαγείας δεν μπορούν να τροποποιηθούν τα πράγματα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί και κάποια νέα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία έχουμε. Αναφέρθηκε και η συγγήτρια σε αυτό, στο EFSD για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Α μην επικεντρώνεται μόνο στα διαθέσιμα μέσα αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αρχίσει να αξιοποιεί περισσότερο και τα επιπλέον χρηματοδοτικά μέσα τα οποία πρόσφατα δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί κάπω, αν θέλετε, και αυτή η ε, πίεση στου υφιστάμενου πόρου. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε η χθεσινή συζήτηση όσον αφορά την πληθώρα αυτή μέσων και είχαμε πει ότι το πιο σημαντικό να δούμε ποιοι είναι οι κοινοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πιο σημαντικό είναι οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί να καταλήξουν σε ένα κοινό όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη στιγμή γίνει αυτό πιστεύω ότι θα βρεθούν και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα. Δίνω πάλι το λόγο, το λόγο τώρα στην εισηγήτρια για να μας συνοψίσει λίγο τα όσα είπε για το έγγραφο αυτοεργασίας που θα οδηγήσει μια έκθεση στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Αρχίζουμε να ξεκαθαρίζουμε κάπως τα πράγματα. Και ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας έδωσε η Επιτροπή και η ΕΤΕ. Με όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα μπω στη δουλειά να ετοιμάσω ένα σχέδιο έκθεσης. Το χρονοδιάγραμμα είναι γνωστό. Το Φεβρουάριος έχει και μια τυρκουάς βδομάδα και μια εβδομάδα στο Στρασβούργο, οπότε δεν έχουμε συνεδρίαση της Επιτροπής μας, δηλαδή είναι πολύ κοντός τελικά ο Φεβρουάριος. Αλλά ίσως θα έπρεπε να ξέρουμε πότε θα έχουμε την επόμενη συνεδρίασή μας και τότε θα φροντίσω να έχω έτοιμο το σχέδιο εκθεσής μου. Όλα οι διαπραγματεύσεις, η συμφωνία πρέπει να έχουν επιτευχθεί για το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο της ΕΤΕ μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές. Σας ευχαριστώ. Και νομίζω ότι η συζήτηση καλύπτει και το Ταμείο Εγγύσεων για τις εξωτερικές δράσεις. Άρα μπορούμε να περάσουμε στην προσεχή έκθεση Ταμείο συνοχή. Χρηματοπιστωτικά μέσα ενισχύσει. Και πάλι εσείς. Ευχαριστώ. Ναι, σήμερα έχω πολλά. Πολύ σύντομα. Πρόκειται για μία γνωμοδότηση που κάνουμε στην Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων που έχει να κάνει με τους σωματοδοτικούς μηχανισμούς και με την πολιτική συνοχής Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε την γνωμοδότησή μας καθαρά στα δημοσιονομικά ζητήματα. Στο πρώτο κομμάτι προσπαθώ να ξεκαθαρίσω ποιος είναι ο ορισμός ή μάλλον ποιος είναι ο στόχος της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων. Γιατί υπάρχουν πολλές αμφιβολίες και ο πειρασμός να πούνε πολλοί ότι αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται για όλα και για τα πάντα. Ενώ θα έπρεπε να τα περιορίσουμε και να ξέρουμε ότι χρησιμοποιούνται εκεί που υπάρχει ένα πρόβλημα στην αγορά ή εκεί όπου οι προϋποθέσεις επενδύσεων δεν είναι οι βέλτιστες. Επίσης, θεώρησα σημαντικό να υπογραμμίσω ότι τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα έχουν την εγγύηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, δηλαδή χρημάτων του Ευρωπαίου Φορολογούμενου, οπότε δεν μπορεί να ασχοληθούμε μόνο με την οικονομική απόδοσή τους, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το στοιχείο ότι πρόκειται για χρήματα δημόσια του κόσμου, εφόσον υπάρχει εγγύηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Και έτσι να το έχουμε υπόψη μας και αυτό το στοιχείο και να προσέχουμε ποιοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι. Τώρα συνοψίζω επίσης τη γνωμοδότησή μου το πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι αυτοί. Αν συγκρίνουμε το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο με αυτό, διαπιστώνουμε ότι διπλασιάστηκε το ποσό στη διάθεση των χρηματοδοτικών αυτών μέσων. Και προσπαθώ να αναφερθώ και στις καθυστερήσεις που καταγγέλουμε εδώ στην Επιτροπή μας για τη λειτουργία όλων των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής ότι δεν γίνονται γρήγορα επενδύσει που χρειάζονται οι περιφερειέ μα γιατί καθυστερούν οι πληρωμέ και τελικά συσσωρεύονται καθυστερήσει απλήρωτοι λογαριασμοί, με δύο λόγια, στο τέλο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Υπογραμμίζω λοιπόν ότι το κοινοβούλιο μας θα πρέπει να ασκεί περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο, να έχει άρα περισσότερες πληροφορίες. Η παρουσίαση τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού και του Omnibus νομίζω ότι θα αποτελέσει μια ευκαιρία για μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες πληροφορίες, πιο εύκολα πρόσβαση σε αυτές και πιο απλούς κανόνες για να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα και επίσης για να συνδυαστεί το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων Juncker με τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ανταλλαγή απόψεων, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο κύριος Νόβακοφ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της, για την πολύ καλή συνεργασία. Νομίζω βρήκαμε ένα καλό πεδίο συνεννόησης, όπου καλύφθηκαν και οι ίσονος σημασίας διαφορές που είχαμε. Φαντάζομαι θα βρεθούν εύκολα συμβαστικές λύσεις. Εγώ έχω και για την Επιτροπή της Περιφερειακής Πολιτικής σχετική έκθεση, καθώς είναι επί της αρμόδια. Θα ήθελα να πω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πρώτη συζήτηση, με το άνοιγμα της συζήτησης για την περίοδο μετά το 2020. Ταυτόχρονα έχουμε το όμνιμπους για το προϋπολογισμό. Έχουμε την ε, ομάδα υψηλού επίπεδου ε, για τους ιδίους σπόρους. Έχουμε την απλούστευση. Άρα λοιπόν είναι η καταλληλότερη στιγμή αυτή για την συζήτηση μιας τέτοιας έκθεσης. Και βέβαια η συμμετοχή των μελών της Επιτροπής των Προπολογισμών έχει κρίσιμη σημασία, γιατί όσο ειδικοί και να είμαστε στο θέμα αυτό, πάντα χρειάζεται να βλέπουμε και την πτυχή του προπολογισμού στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής έχω ένα συνάδελφο που λέει καλύτερη προετοιμασία, ίσον καλύτερα αποτελέσματα. Ε, αυτό λέω και εγώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως είπα και στη Ρέτζη, εάν θεωρήσουμε ότι χρηματοδοτικά μέσα και δάνεια είναι δύο μηχανές του αυτού αεροπλάνου, δεν μπορούμε να έχουμε ένα αεροπλάνο το οποίο θα κινηθεί και θα απογειωθεί με ένα μόνο κινητήρα εν λειτουργία. Χρειάζονται λοιπόν και οι δύο πτυχές πρέπει να λειτουργήσουν καλά και νομίζω ότι αυτή η έκθεση και η γνωμοδότηση θα αποτελέσουν ορόσημο για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε κάποιον άλλον. Κυρία Καρδιά Σαβάλα, όχι, για να διευκρινίσετε τίποτα κλείνουμε. Η τροπολογίε το αργότερο 31 Ιανουαρίου στις 12 για την Επιτροπή των Προϋπολογισμών η γνωμοδότηση ψηφίστε στους προϋπολογισμούς 6 Μαρτίου. Γνωμοδότηση υπενθυμίζω. Η επίτηση της επιτροπή είναι η περιφερειακή και ψηφίζει στις 20 Μαρτίου. Και τώρα... Ο κύριος Κορσάλης Πόνς. Διαχείριση αλλιευτικών στόλων στις εξόχως αποκέντρες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με την γνωμοδότηση αυτή θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη στην πραγματική κατάσταση των ελευτικών σκαφών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες προκειμένου να προτείνει ενισχύσεις για τους ελευτικούς αυτούς στόλους. Πρόκειται μόνο, επιμένω, για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Είναι μια εκδίκηση των περιφερειών αυτών όπου ο τοπικός ε, αλληλευτικός στόλος έχει γεράσει πάρα πολύ και τίθεται και θέμα και ασφάλειας, όχι μόνο άνεσης πάνω στα σκάφη αυτά. Προ το παρόν δεν υπάρχουν ενισχύσει για την ανανέωση των σκαφών αυτών. Καταργήθηκαν με τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική το 2002, προκειμένου να μην υπάρξει υπερβολικά μεγάλη αλληλευτική ικανότητα, η οποία στο παρελθόν οδήγησε σε υπερεκμετάλλευση των αλληλευτικών πόρων. Όμω, πρέπει να σα πω εδώ ότι οι εξόχω απόκεντρε περιφέρειες, εξόχω απόκεντρε περιφέρειες επαναλαμβάνω, διαθέτουν μικρής κλίμακας αλλιευτικό στόλο. Δεν ε, κάνει ζημιά στο περιβάλλον. Χρησιμοποιούν παραδοσιακούς τρόπους αλίας. Οπότε θα έπρεπε να μπορούν να υπάρχουν τέτοιες ανισχύσεις. Είναι το άρθρο 349 τη Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση που προτείνει ειδικά μέτρα για τι περιοχέ αυτέ, ακριβώ επειδή κοινωνικά, ε, οικονομικά αλλά και γεωγραφικά έχουν μια ιδιαίτερη κατάσταση. Πρέπει να ξέρουμε ότι η κρίση έπληξε ακόμα περισσότερο τι περιφέρειες αυτέ, που έχουν και ανεργία παραπάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Γι' αυτό και ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες μέλη να απλοποιήσουν την πρόσβαση και την χρήση των διαρθρωτικών ταμείων ή και άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς προκειμένου να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών που βρίσκονται τόσο μακριά από το κέντρο της Ευρώπης. 30 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και κατά τα άλλα είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι παρατηρήσεις έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Ε, η κυρία Ζαμπάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεση αυτή δεν είναι δικιά μου. Η κυρία Τωμά όμως δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, οπότε έχω κάποια σχόλια. Ε, συμφωνούμε, είμαστε σαφώς υπέρ των ενισχύσεων αυτών για την ανανέωση των ελευτικών σκόλων, γιατί όπως έλεγε και ο κ. Πόνς, είναι παραδοσιακά σκάφη μικρής κλίμακα οπότε δεν κάνουν ζημιά στο περιβάλλον. Αλλά μια που εμεί είμαστε προπολογισμού, πρέπει να δούμε τι δημοσιονομικές επιπτώσεις έχει αυτό. Από την άλλη, πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε ένα καθεστώς ε, ποσέ για παράδειγμα για την Αλία όπως υπάρχει για τη Γεωργία και θα μπορούσε να είναι μια καλή πρόταση αυτή. Τίποτα άλλο. Εννοείται θα υποβάλουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και σίγουρα θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Πρόεδρος, ωραία. Πολλά υποσχόμενα όλα αυτά. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Οπότε ο εισηγητή μα μας είπε ότι οι τροπολογίε πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο στι 12 το μεσημέρι στι 30 Ιανουαρίου. Θα ψηφίσουμε στι 6 Μαρτίου στην Επιτροπή μα και στην αρμόδια επί της ουσίας ε, Επιτροπή στις 20 Μαρτίου, στην Επιτροπή Αλίας. Αυτά. Σας προτείνω. Δεν έχω τίποτα άλλο. 9 Φεβρουαρίου είναι η προσοχή συνεδρία τη Επιτροπή των Προπολογισμών εδώ στι Βρυξέλλε. Έχετε την ενημέρωση για τα υπόλοιπα προ εκαθάριση, ραλ, προ ρευστοποίηση. Ε, ζητεί κανεί άλλο το λόγο. Όχι. Κύριε λοιπόν, το πέρασε τη συνεδριά σα. Στι 10.30 ξεκινούμε του συντονιστέ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.